Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε, διότι πρέπει να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ καθίστε. E λοιπόν, περνάμε μέσα στην ψηφοφορία. Τη μία και μοναδική που έχουμε για σήμερα για την έκθεση της κυρίας Μαρίας ε, Μιούνις Δερκουρκίσα με τίτλο Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος φορέας, ο ρόλος της εις πολυμερής οργανώσης». Καλώς. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική υπαριθμό 5. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ, τη συμβαστική τροπολογία 5 κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε μέσω στην τροπολογία 62, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση, η οποία και αρχίζει. Ηλεκτρονική. Ηλεκτρονική επί της 72. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ε, la votazione. Πέρας. Όχι, άμεση, με συγχωρείτε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, εντάξει. Ας περιμένουμε, ας περιμένουμε. Με την άνεσή σας. Ci sono 50 schede inserite. Παρακαλώ βάλτε τις κάρτες σας και ψηφίστε. 52 ψηφίσαντες. 27 έναντι 23 εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε. Εγκρίθηκε η 72, ψηφίζουμε την 74. 74. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ας ε, περιμένουμε τον κύριο Μπρόκ να τελειώσει την τηλεφωνική του συνομιλία για να μην τον ενοχλούμε. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82. Αν θέλετε να ελέγξουμε. Αρχίζει η ηλεκτρονική επί της τροπολογίας 81. 54-54. 54 54 Όχι. Απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 7. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές, αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του δεύτερου τμήματος του συμβιβασμού 7. 54 ψηφίσαντες απορρίπτεται για δύο ψήφους. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86. 86 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές Αποχές δεν είναι σαφές. 90. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. «55 για μία ψήφο απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Ωραία. Ελέγχουμε την 91. 91. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Λείπει μία ψήφος. Κάποιος είναι αφηρημένος. Τι να κάνουμε. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αποσύρεται η 93, ψηφίζουμε την 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά 101 αρχίζει η ψηφοφορία 58 ψηφίσαντες, 31 ε, κατά, 25 υπέρ. Απορρίπτεται, 102 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται, 103. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε, επί της 102 αρχίζει η ηλεκτρονική. 58 ψηφίσαντες, ε, απορρίπτεται, 32 κατά, έναντι 25, 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 αρχίζει ηλεκτρονική ηλεκτρονικός έλεγχος 104 58 ψηφίσαντες, ισοψηφία απορρίπτεται. Είχατε δίκιο να αμφισβητήσετε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν ε, περνά λόγω ισοψηφία. 8. Συμβασμός 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 120 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αποσύρεται 122, 125. Α, εντάξει, 121 Αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία, αφού θέλετε έλεγχο. 121. Ηλεκτρονικός έλεγχος, πέρας. 56 ε, έναντι 2. Δεν πρέπει να αλλάξω γυαλιά. Μου το επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα. Αποσύρεται 122-125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 με την προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε δεν είναι σαφές. 130. Αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επί της 130. 130 για τους αφηρημένους. Δύο δεν ψήφισαν. Α, τώρα ψήφισαν. 21 υπέρ, 31 κατά. 131. Α, καταπίπτει 131. Γιατί εγκρίθηκε η 129 και απορρίφθηκε 130. Περνάμε, περνάμε τώρα στην 132. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μάλλον με συγχωρείτε. Διανατάσεως υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται, μου φαίνεται. Αλλά αν θέλετε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά προφορική 2. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Είχετε δίκιο, εγκρίθηκε για μία ψήφο. Άρα τώρα περνάμε στην 137 υπέρ της 137. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. 137 αρχίζει η ψηφοφορία. Δύο συναδελφοί δεν ψήφισαν. Ένας τώρα. Ένας ξεχάστηκε. Ωραία ψήφισε. Πέρασε. 28 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Αποσύρεται 139, 140 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 10 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 150. 149. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 149. Ψήφισαν όλοι πέρας. 29-28 το απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές ε, μου φαίνεται ότι απορρίπτεται 152 εντάξει 151 ηλεκτρονικός έλεγχος δεν πρέπει ποτέ να λέω μου φαίνεται 59 ψήφισαν. Απορρίφθηκε. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε την 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε. Αρχίζει ο έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος επί της 14. Τρεις δεν ψήφισαν, δύο τώρα, δύο συνάδελφοι δεν ψήφισαν. Πέρας, 34 υπέρ, 22 κατά εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Αρχίζει ηλεκτρονική. Επί της 15. 15. Δύο δεν ψήφισαν. Πέρας. 28 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. 16. 16 με συγχωρείτε. Και εδώ δεν είναι σαφές. 16. 16. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της 16. Πέρας. Εγκρίνεται με 33 ψήφους. 17. 17 τώρα. 17. Υπέρ. Ψηφίζουμε την 17. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Πείτε. Ποιο, τι ψηφίζουμε. Γιατί εδώ έχουμε διαφορετικούς, διαφορετική αρρύθμιση. Είδαμε τον πίνακα και μιλούσαμε και μεταξύ μας βέβαια. 17 και η προηγούμενη και θεωρήσαμε ότι ήταν η 17. Μπορούμε να ξαναψηφίσουμε την 16. Eh, eh, Με συγχωρείτε. Μα, είπα 16, εγώ είπα 16. Τότε ήταν λάθος επί της οθόνης. Mm. Θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός να ακούς τη φωνή του Προέδρου, την προεδρική φωνή, η που υπερέχει. Δεν μπορεί να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Λυπάμαι. 17 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 17. Αρχίζει η ψηφοφορία. 17, 17. Μην κοιτάτε την οθόνη. Σα είπα. Ψηφίζουμε τη 17. Δύο δεν ψήφισαν, αλλά τελειώνουμε. Πέρας. Για μία ψήφο απορρίπτεται. 18 υπέρ. 18 τώρα υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Συμβιβασμό 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά δεν είναι σαφές. Αρχίζουμε την ηλεκτρονική. 27. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 32 κατά, 25 υπέρ. Απορρίπτεται. Πάμε στην 20... Πάμε στην 30. 30. Υπέρ της 30. Κατά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 αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές ε, δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε επί τη 40. Ελέγχουμε την 40. Πέρας. Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 30-30. Απορρίπτεται. 41. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε 46. Ελέγχουμε την 46. Αρχίζει ηλεκτρονική. Πέρασε, ψήφισαν όλοι 29 κατά, 31 υπέρ, εγκρίνεται 4 υπέρ της τροπολογίας συμβάσμου 4. Κατά. Δεν σηκώσα τα χέρια. Άρα νομίζω ότι είμαστε υπέρ 53.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 αποχές απορρίπτεται Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Υπάρχει μια πρόταση λειτουργικής φύσης ε, να ψηφίσουμε μπλοκ από την 4 έως την 10. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτή την επιτάχυνση, όχι? Μάλι, va bene. Ωραία. Πέντε, μία-μία. Με συγχωρείτε, 4, 4. Ψηφίζουμε την ίντα 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 11. Ωραία, αρχίζει η ηλεκτρονική επί της 11. 60 ψηφίσαντες, 27 υπέρ, 33 κατά απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στην έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί, αρχίζει ηλεκτρονική. Δεν έχουν ψηφίσει δύο συνάδελφοι. Πέρας, παρόλα αυτά. Ένας λείπει, αλλά κλείνουμε.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 Διακόπτω καμιά ιδιωτική συζήτηση. Κύριε Μπροκ, δεν είχατε ζητήσει το λόγο. Πάρτε μαζί την ε, κάρτα σας, αλλιώς θα την ξεχάσετε. Και θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την ακρόαση για την ε, κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο, Τουρκμενιστάν, ανταλλαγή απόψεων με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Λίγα λεπτά διακοπή. Onorevole Salafranca, prego. Eh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, συγγήτρια για την έγκριση της έκθεσής της και το αποτέλεσμα αυτής και ήθελα παρακαλώ να ζητήσω να γραφεί στα πρακτικά. Έλεγα κύριε Πρόεδρε ότι Συγχαίρω την εισηγήτρια για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αλλά θα ήθελα εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας να γραφεί στα πρακτικά, γιατί αυτά τα πράγματα καλό είναι να λέγονται. Ότι, παρά το γεγονός ότι η ίδια κατέβασε ε, διάφορες προφορικές τροπολογίες, η δική μου πολιτική ομάδα την υποστήριξε. Θυμίζω ότι η εισηγήτρια επανειλημμένα χαρακτηρίστηκε ε, από την απόρριψη της ε, ορισμένων ε, και πολλών προφορικών τροπολογιών που είχε καταθέσει η δική μου πολιτική ομάδα. Σας ευχαριστώ για αυτή τη διευκρίνηση. Περνάμε τώρα στο σημείο 8 που όπως σας είπα αφορά μια ανταλλαγή απόψεων με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Γνωρίζετε ότι η εταιρική συμφωνία και συμφωνία συνεργασίας που εγκρίθηκε και που μάλλον θα πρέπει να εγκριθεί, θα εγκριθεί την 1η Ιουνίου, έθεσε στο επίκεντρο των εργασιών μας το θέμα αυτό. Τις χώρες δηλαδή που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή του κόσμου και ιδιαίτερα το Τουρκμενιστάν που γνωρίζουν μεγάλη αστάθεια, κυβερνητική αστάθεια και δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, όπως έχουμε μάθει εμείς και όπως τις γνωρίζουμε εμείς. Και οι σχέσεις μας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας προβλέπει μια τέτοια ανταλλαγή απόψεων. Προβλέπεται λοιπόν μία επίσκεψη από τις 26 έως 30 Απριλίου στο Τουρκμενιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Επειδή ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθουμε σε επαφή με ανεξάρτητες οργανώσεις, ιδιαίτερα στο Τουρκμενιστάν, κρίναμε σκόπιμο να τις συναντήσουμε εδώ, στο δικό μας περιβάλλον, για να μπορέσουμε να ακούσουμε την άποψη, μια μη κυβερνητική άποψη που θα μας διαφωτίσει. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φαρίτ Τουκμπατουλίν, ο οποίος είναι ένας ακτιβιστής που ε, έχει ε, διωχθεί από την κυβέρνησή του και ακόμα και στην εξορία του στην Ευρώπη βρίσκεται σε επαφή με τους συμπατριώτες του και γνωρίζει την κατάσταση από την πηγή. Και ο κύριος Γιάσης Μάβεντοφ είναι ένας εκπρόσωπος ε, μιας ε, πολιτικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κυρία Σβέντεν Γκόλστον που είναι εκπρόσωπος του Human Rights Watch, μια οργάνωση που γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που στο παρελθόν ε, ακούστηκε, εισακούστηκε η άποψή της ε, στη, εδώ στο σώμα μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Χάουταλα, η οποία είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κυρία Χάουταλα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το υπόβαθρο αυτής της συζήτησης είναι το εξής. Η Επιτροπή Εξωτερικών Θέσεων υιοθέτησε το Φεβρουάριο ένα ψήφισμα μη νομοθετικό, η οποία είναι κρίσιμη, διότι αναφέρεται στις προϋποθέσεις ε, για την επικύρωση της, συμφωνία, της εταιρικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκμενιστάν. Όπως είπα δεν είναι νομοθετικό, ε, ε, δεν έχει νομοθετικής φύσης και ε, το ψήφισμα αυτό και το συμπέρασμα τότε της συζήτησης ήταν ότι η τελική ψηφοφορία του Κοινοβουλίου μέσα στα πλαίσια του Συμφωνίας Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης θα ε, γίνει μετά από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας ε, και στην συνεπιτοπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτή η επίσκεψη τώρα θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και επίσης η επίσκεψη το Τουρκμενιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Αυτή είναι μία, ε, ένα παράδειγμα μία υπόθεσης ε, την οποία, η οποία μπορεί να δείξει την ε, θέση του Κοινοβουλίου σε αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας και εταιρική σχέσης επί τη βάση της συνθήκης της Λισαβόνας. Το Κοινοβούλιο έχει τώρα τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να ε, μην εγκρίνει Διεθνή συμφωνίες με τη βοήθεια της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και ε, την ε, εισηγείται κυρία Νίκολάη. Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζήτησε τις πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής. Η εικόνα συνάδει με αυτά τα οποία αναφέρει το μη θετικό ψήφισμα που και στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν ένα άλλο διαθεσμικό θέμα, το, το μη δημοθετικό ψήφισμα, το ε, Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί ε, την εφαρμογή, ζητάει την εφαρμογή ορισμένων ε, εποπτικών δράσεων, δηλαδή ζητάει την παρακολούθηση ορισμένων ενεργειών. Ε, μία ερώτηση στην ε, η υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας δηλαδή, και η απάντηση ήταν πάρα πολύ απογοητευτική. Η Ευρωπαϊκή <clears throat> Υπηρεσία Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας είπε ότι δεν θα δώσει συνέχεια σε αυτό το ψήφισμα διαβουλεύτηκε ε, με νομικούς εμπειρογνώμενους και είπε ότι ένας τέτοιος μηχανισμός εποπτείας και παρακολούθησης θα διαταράξει τη δυσορροπία ε, των σχέσεων. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθήσει από πολύ κοντά την εξέλιξη, διότι είναι δική μας αρμοδιότητα. Και προτείνω, Πρόεδρε, εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων να ζητήσετε μία νομική γνωμοδότηση για να δούμε εάν η γνωμοδότηση της υπηρεσία ε, ε, ε, εξωτερικής πολιτικής είναι σωστή. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πρέπει να ζητήσει από τη δική του την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκδώσει μια γνωμοδότηση, διότι σας είπα, εδώ πρόκειται για την, το δικαίωμα που έχουμε να παρακολουθούμε την υλοποίηση των συμφωνιών ε, συνεργασίες και εταιρικής σχέσης. Ε, άρα λοιπόν ε, πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν και αυτό είναι το υπόβαθρο της συζήτησης που είχαμε στην υποεπιτροπή μας. Ευχαριστώ την Πρόεδρο Χάουταλα. Περνάμε τώρα στην ακρόαση αρχίζοντας με τον κύριο Φαρίτ Τουκμπατουλίν στον οποίο θα δώσω το λόγο και θα ήθελα να λάβει το λόγο για πέντε λεπτά. Θερμή παράκληση έτσι ώστε να υπάρξει διάλογος, να έχουμε διάλογο με τους συναδέλφους. Έχετε το λόγο, κύριε του Ευχαριστώ Спасибо большое э, за приглашение на столь важное для нас мероприятие и я был рад услышать э, о том, что все-таки э, представители э, Европейского парламента интересуются ситуацией в Туркменистане. Καλημέρα σας. Είμαι πολύ ευτυχής που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται έντονη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν. Είμαι ευτυχής που διαπιστώνω το ενδιαφέρον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μου. Τα τελευταία 20 χρόνια στο Τουρκμενιστάν υπάρχει ένα απολυταρχικό καθεστώς ε, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί από πολλούς διεθνείς οργανισμούς ε, παρόλο που αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί όπως η ΟΑΣΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι μας λένε ότι παρόλο το καθεστώς αυτό υπάρχει ένας διάλογος και ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. Ο προηγούμενος πρόεδρος παρετήθηκε, αλλά ο νυν πρόεδρος ακολουθεί ακριβώς την ίδια πολιτική. Όταν στο Τουρκμενιστάν υιοθετείται κάποιο νομοσχέδιο. Ορισμένα από αυτά είναι ε, καλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διορθώνεται όλη η κατάσταση, διότι ο τρόπος ε, εφαρμογής της νομοθεσίας είναι πολύ διαφορετικός. Ναι, μεν καλά επικυρώνεται ή υιοθετείται ένα νομοθετικό ε, μέσον, αλλά εν συνεχεία δεν εφαρμόζεται. Γι' αυτό θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Η πολιτική ε, τιμωρίας, ε, εγκλισμού πολιτών σε ψυχιατρικά νοσοκομεία έχει αναζωογονηθεί και εφαρμόζεται ξανά. Υπάρχουν πολλοί πολίτες που χωρίς λόγο υποχρεώνονται να κλειστούν σε ψυχιατρικά ιδρύματα και το Μάρτιο ο Αμάγγελ που είναι 80 χρονών ο άνθρωπος ε, αλλά τόλμησε να δώσει μία συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Liberty, Ελευθερία ε, κλείστηκε σε ψυχιατρίο. Ένας δημοσιογράφος του ίδιου ραδιοφωνικού σταθμού ε, τον παρακολουθούσε η μυστική αστυνομία και τιμωρήθηκε, διώχτηκε πολλές φορές το όνομά του είναι στη μαύρη λίστα και δεν μπορεί να εργαστεί στο Τουρκμενιστάν ούτε μπορεί να φύγει από τη χώρα αλλά και ο γιος του δεν μπορεί να βρει δουλειά και να φύγει από το Τουρκμενιστάν ο γιος του μετά από αυτή την κατάσταση αυτοκτόνησε και στο τέλος του 2010 το Δεκέμβριο το πετροβολήθηκε το, το σπίτι ενός άλλου πολίτη από μία ομάδα υποτίθεται αλητών και ε, υπάρχει άλλη μια τραγωδία στην οικογένεια Μπερντίεφ αυτή η οικογένεια ήταν επιχειρηματίες και η μυστική αστυνομία κατάσχεσε όλα τους, όλη τους την ιδιοκτησία, τους ε, συνέλαβε, βασανίστηκαν ε, τους ε, έσυρε στα δικαστήρια όπου δεν τους απαγγέλθηκε κατηγορητήριο. Εν πάση περιπτώσει άσκησε τρομακτική πίεση πάνω στα μέλη της οικογένειας και η μητέρα η Ατσέμπαλ ε, κλείστηκε πολλές φορές στο ψυχιατρίο. Η γυναίκα προσπάθησε επανειλημμένως να αυτοκτονήσει. ο Αχμεντανάιεφ προσπάθησε να διαφύγει στη Μόσχα διότι χρειαζόταν ιατρική θεραπεία όμως ποτέ δεν μπόρεσε να φύγει από το Τουρκμενιστάν όπου δεν μπορούσε να έχει την περίθαλψη που χρειαζόταν διότι ήταν μέλος της αντιπολίτευσης. Ε, αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι συλλαμβάνονται μέλη της οικογένειας και κρατούνται ως όμοιροι των ε, ως όμοιροι μέλη της οικογένειας αντιπολιτευομένων ατόμων. Έχω και άλλα παραδείγματα ε, πρόσφατα. Ε, μία ομάδα νέων τραγουδιστών συνελήφθησαν διότι προσπάθησαν να δώσουν μία συνέντευξη στο τουρκικό ραδιόφωνο αλλά και συγγενείς αυτών των νέων παιδιών της ε, ομάδας αυτής συνελήφθησαν και πιέστηκαν. Ε, ξέρω ότι έχουμε πάρα πολύ λίγο καιρό και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. E σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να προωθήσουμε έμπρακτα έναν διάλογο μετά από την εισήγησή σας. Ο κύριος Γιάννης Λαφμάμεντοφ, που είναι ο ε, εκπρόσωπος της Δημοκρατικής οργάνωσης πολιτών από το Τουρκμενιστάν. Σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά επίσης για να έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε αυτόν τον διάλογο που επιθυμούμε στη συνέχεια. Έχετε το λόγο. У меня появилась возможность выступить перед вами с этой высокой трибуны. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να παρέμβω και να πω ότι όταν ε, συζητάτε τη σχέση σας με το Τουρκμενιστάν να μην κάνετε λάθη τα οποία είχαν ε, διαπράξει συνάδελφοι από τα Ηνωμένα Έθνη, διότι δεν εξέτασαν την κατάσταση εις βάθος και δεν ζήτησαν από την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Βεβαίως ε, υποστηρίχθηκε η ουδετερότητα του Τουρκμενιστάν, αλλά το Τουρκμενιστάν ποτέ ε, δεν ε, μπόρεσε να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις του. Γι' αυτό όταν συζητάτε για θέματα που αφορούν το Τουρκμενιστάν και λαμβάνετε αποφάσεις, να το λαμβάνετε αυτό σοβαρά υπόψη. Είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστείτε με κυβερνήσεις και με κατασταλτικά καθεστώτα. Θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν. Ε, δυστυχώς οι επικεφαλής είναι πολύ οξυδερκείς και ξέρουν πολύ καλά πώς μπορούν να παρακάμψουν τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους. Νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να ζητήσουμε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και να δοθεί τέλος σε αυτό το καθεστώς καταστολής. 15.000 ε, άνθρωποι θα πρέπει να βγουν από τη μαύρη λίστα και θα πρέπει να επαναδιαρθρώσουμε την κοινωνία των πολιτών. Εάν τηρηθούν αυτοί οι όροι, δεν θα υπάρχει κανένα πρόσκομα για μελλοντική συνεργασία ως προς την εμπορική εταιρική σχέση. Και θα ήθελα να σας επισύρω επίσης την προσοχή στο εξής γεγονός. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια φυλακή Αντελάντου Μπέ η οποία μοιάζει με στρατόπεδο συγκέντρωσης και περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Θα ήθελα να σας πω ότι οι φυλακισμένοι, οι κρατούμενοι, δεν μπορούν να συναντηθούν με τους συγγενείς τους και δεν έχουν δικαίωμα να συναντηθούν με τους συνηγόρους τους. Άρα είναι σαν να βρίσκονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, χωρίς κανένα δικαίωμα. Θα ήθελα να το συζητήσω συζητήσετε το θέμα αυτής της συγκεκριμένης φυλακής με την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν. Ξέρω ότι δεν διαθέτουμε πολύ χρόνο και θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να συζητήσετε αυτή την κατάσταση με τις μητέρες υγιή των οποίων κρατούνται σε πολλές φυλακές. Επίσης νέοι οι οποίοι είναι ναρκωμανείς και δυστυχώς ε, καταναγκάστηκαν στο να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε ότι τα ναρκωτικά έρχονται από το Τατζικιστάν σε μεγάλες ποσότητες και η κυβέρνηση φαίνεται σαν να προωθεί αυτό το εμπόριο. Και επειδή οι διεθνείς οργανισμοί ακολουθούν παθητική στάση, και είναι σιωπηρή, η σιωπή σημαίνει και αποδοχή. Αποδοχή των πράξεων της κυβέρνησής μας. Θα ήθελα λοιπόν να θέσετε ορισμένους προκαταρκτικούς όρους και μετά να αποφασίσετε αν μπορείτε να συνεργαστείτε με το Τουρκμενιστάν. Ε, δεν θα πρέπει να υποστηρίξετε τις ε, οικονομικές σχέσεις κατά της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να βάζουμε την, ε, σε παρασετιώδη συνάφεια τη δημοκρατία με την οικονομία. Διαφορετικά είναι σαν να έχουμε να κάνουμε με ένα κρυφό λόμπι των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Το Τουρκμενιστάν προωθεί τα αποθέματα του κατά 2-3% στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει και αυτό να λάβετε υπόψη σοβαρά στις συζητήσεις σας. Ευχαριστούμε κύριο ε, Μάβεντοφ, η κυρία Βερονίκ Τζένκιν Γκόλστον έχει το λόγο που είναι εκπρόσωπος της οργάνωσης Human Rights Watch που γνωρίζουμε διότι ήδη έχει παρέμβει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν και για τη δραστηριότητα του καθεστώτος σε διάφορους οργανισμούς της διεθνούς κοινότητας. Έχετε το λόγο. Και όπως είπα και για τους άλλους παρεμβαίνοντες, θα ήθελα να αρκεστείτε στα πέντε λεπτά ή δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη. Κύριοι βουλευτές, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας ε, σε ένα έγγραφο που έχουμε εκπονήσει από τη Human Rights Watch για το Τουρκμενιστάν εν ώψη της ε, ενασχόλησής σας ε, με τη χώρα αυτή. Ε, ο χρόνος μου είναι πολύτιμος εδώ και δεν θα σας δώσω επισκόπηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επειδή έχετε το κείμενο και μεταξύ άλλων τα πάρα πολύ δυνατές συμμαρτυρίες που ακούσατε μόλις για το πώς έχει η κατάσταση στη χώρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λοιπόν αβυσαλαία η κατάσταση αυτή και θα προσπαθήσω να τη συνδέσω με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Τουρκμενιστάν και σε σχέση με το όσα είπε η κυρία Χάουτα, αλλά πολύ σημαντικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλέον έχει μια θαυμάσια ευκαιρία να εξασφαλίσει ε, ότι θα διαδραματίσει το πρωταγωνιστικό του ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και θα το συνδέσει με τις βελτιώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι συμβαίνει ακριβώς. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με ένα από τα πιο κατασταλτικά καθεστώτα παγκοσμίω, χωρίς να απαιτήσει βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αντάλλαγμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα είναι ε, το μόνο θεσμικό ε, όργανο που θέλει ε, να βάλει ορόσημα και στοιχεία benchmarks για αξιολόγηση των συμφωνιών εταιρική σχέση, συνεργασία και δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι δεν είναι γεγονός αυτό στη συμφωνία σήμερα. Παρόλο που το 2009 ενέκρινε τη συμφωνία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε έναυσμα και κίνητρο για μεταρρύθμιση, αλλά αυτή η μεταρρύθμιση δεν επήλθε. Και Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υποσχέθηκαν στο Κοινοβούλιο ότι θα το παρακολουθούν ε, αυτό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μελήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δρόμο προς ε, τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, PCA. Ε, δεν έγινε όμω τίποτα τέτοιο από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Τι συμβαίνει εδώ λοιπόν. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έδειξε την παραμικρή προθυμία να μεταρρυθμίσει και από την άλλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει καταβάλει μια πραγματική προσπάθεια να πιέσει προ την κατεύθυνση αυτή. Παρ' όλα αυτά το ψήφισμα όπω εγκρίθηκε στην Επιτροπή σα νωρίτερα φέτο ενέκρινε τη Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία. Ε, με ένα μηχανισμό συνοδευτικό για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όπως είπε η κυρία Χάουταλα, η ε, Υπηρεσία Εξωτερικής δράση ξεκαθάρισε στη συνέχεια ότι ο μηχανισμό δεν πρόκειται να υπάρξει. Και αυτό το επιβεβαίωσε και άλλος εκπρόσωπος τη ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση στην εξωτερική υπηρεσία λοιπόν στη χθεσινή συνεδρίαση τη αντιπροσωπεία με την Κεντρική Ασία. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει, απέτυχε να απαντήσει ε, στο επίσης κομβικό και βασικό ερώτημα και αίτημα που ήταν μια μελέτη αντικτύπου που είχε η προηγούμενη συμφωνία με τον Τουρκμενιστάν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διεθνής Εμπορική Συμφωνία. Και ε, βασιζόταν ε, στην ελπίδα ότι θα βελτιωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η επικείμενη λοιπόν επίσκεψή σας είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την αξιολόγηση και εκτίμηση της κατάστασης που παραμένει ικτρή και θα πρέπει να σκεφτούν ε, οι αρχές της χώρας και να αποδείξουν ότι είναι πρόθυμες να κάνουν μεταρρυθμίσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει ε, όπως λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά τις αλλαγές γιατί τέτοια ε, σημεία δεν υπάρχουν και τέτοιες ενδείξεις. Θα πρέπει να διδαχθούμε ε, από άλλα μέρη του κόσμου και μεταξύ άλλων την ε, Μέση Ανατολή και πώς μπορούμε να ε, δράσουμε και στη χώρα αυτή. Είναι μεγάλες οι ομοιότητες και θα πρέπει να αναθεωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναθεωρεί και τώρα κάποιες παρανοήσεις και λανθασμένες στη Μέση Ανατολή, αλλά θα πρέπει αυτό να επεκταθεί και σε άλλε περιοχέ και σε άλλε κυβερνήσει και στο Τουρκμενιστάν, όπου υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα που επικρατούν εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είτε αυτά είναι ε, οικονομικά, ασφαλεία είτε άλλα. Αυτά τα δύο δεν είναι αλληλοαποκλείωμενα όμω. Χθε στη συνεδρίαση τη Αντιπροσωπεία για την Κεντρική ε, Ασία, η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είπε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω. Γιατί καταρρύπτει ε, το επιχείρημα κατά της ε, πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λέει ότι έδειξε ειλικρινή προθυμία να ε, εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τουρκμενιστάν, χωρίς να θέλει να περιορίσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα. Είναι μια σχέση που θέλει και η τουρκμενική κυβέρνηση, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η Ένωση έχει ε, μέσα για να πιέσει και θα πρέπει να τα αξιοποιήσει πλήρως. Πώς θα τα αξιοποιήσει πλήρως, τι σημαίνει αυτό. Να μην τους δώσουμε δωρεάν τη Συμφωνία εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας. Να είναι πραγματικά ένα όχημα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή η συμφωνία. Και θα πρέπει να επιμείνει η Ένωση να βελτιωθεί η κατάσταση πριν ε, υπογραφεί η συμφωνία. Ευχαριστούμε την κυρία Γκόλστον. Τελειώσατε. <laughs> Άμεση Όχι ακριβώς. Με συγχωρείτε, ίσως μπορέσετε να απαντήσετε μετά. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα δώσω το λόγο στην κυρία Φυσέρα από την ΕΙΕΔ που ίσως έχει κάτι να προσθέσει σε σχέση με την όλη πλαισίωση του ζητήματο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας. Λίγα λόγια μόνο θα πω επειδή μας πιέζει και ο χρόνος. Θα ήθελα να αρχίσω εκφράζοντας την εκτίμησή μου για τις ε, παρεμβάσεις τις οποίες άκουσα από τους προλαλήσαντες. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο που κάνουν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί στην περιφέρεια και στη χώρα και ε, κατανοούμε ότι είναι μια τεράστια πρόκληση. Συμφωνώ απόλυτα ότι η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν δημιουργεί μεγάλες επιφυλάξεις και ανησυχίες ε, όπως και σε άλλες χώρες στην Κεντρική Ασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως επίκεντρο στις σχέσεις με τις χώρες αυτές και έχει εκπονήσει μια στρατηγική η οποία εγκρίθηκε, υιοθετήθηκε το 2007. Από τότε έχουμε έναν τακτικό ετήσιο διάλογο με κάθε μία από τις χώρες αυτές συμπεριλαμβανομένου και του Τουρκμενιστάν. Είναι συζητήσεις δύσκολες αλλά γίνονται με αμεσότητα και υπευθυνότητα. Και έτσι μπορούμε να συζητήσουμε με διάφορους εκπροσώπους του Τουρκμενιστάν. Μέσα στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού έχουμε αναπτύξει, αναπτύξει επίσης ένα διάλογο με την ε, κοινωνία ε, των πολιτών ε, και με άλλους ενδιαφερόμενους η σχέση των, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο διάλογο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα αυτό, ούτε μόνο με εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων. Πρόσφατα συνεδριάσαμε στο, τα, στην Τασκένδη και συζητήσαμε μία σειρά θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που ανησυχούν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι χώρες όπως το Τουρκμενιστάν και εδώ πάλι τονίζω ότι συμφωνώ πολύ με αυτά που ελέγχθησαν σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύουμε λοιπόν στο διάλογο, στη συζήτηση και δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτύχουμε πρόοδο βραχυπρόθεσμα. Είναι μία μακροπρόθεσμη προσπάθεια. Όσο πιο πολύ Είμαστε σε επαφή, τόσο πιο πολύ μπορούμε να πιέσουμε και να ενσαρρύνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το PCA θα μας δώσει τη δυνατότητα νέων μέσων ε, περαιτέρω συνεργασίας και θα δημιουργήσει και μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία θα διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων. Αυτή η συμφωνία λοιπόν ε, εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ε, περιλαμβάνει και το θέμα του εποπτικού μηχανισμού δεν θα σταθώ σε αυτό, αλλά οπωσδήποτε η συμφωνία αυτή θα μας δώσει μια σωστή βάση επαφών ε, με όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Καταλήγοντας θέλω να τονίσω το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ε, με μεγάλη ανακούφιση ακούσαμε ότι θα γίνει η επίσκεψη της αντιπροσωπείας στο Τουρκμενιστάν και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για το τι θα διαπιστώσετε εκεί. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους προσωπικά ε, τους ε, συμμετέχοντες σήμερα στη συζήτηση αυτή και προσβλέπουμε μεγάλη ικανοποίηση στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πέτερινγκ, πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να εκφράσω την εκτίμησή μου και για τον Φαρίντε του Κμπάτουλιν και για τον ε, Νάμπιτοφ και την Βερόνικα Τσέντερ Γκόλστον από τη Σουηδία, την καλεσμένη μας, όλους τους καλεσμένους μας ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Τουκμπατουλίν μπόρεσε να εγκατασταθεί στην ε, Αυστρία και ο κύριος Νεμπάτοφ στην ε, Ολλανδία. Ξέρουμε τι, τα αισθήματα των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και να ζητήσουν άσυλο σε άλλες χώρες. Θέλω να αφαιρθώ στο θέμα της σταθερότητας. Σε εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά στην διεθνή σφαίρα πολλές φορές ακούγεται η έννοια σταθερότητα, σταθερότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ελευθερία ελευθερία και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Ήδη στο επικομμουνιστικό καθεστώτων η σταθερότητα ήταν μια εσφαλμένη αντίληψη διότι απέβαινε εις βάρος των ανθρώπων που έπρεπε και ήθελαν να ζήσουν ελεύθερα. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε σταθερότητα τα, καλύπτονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο, το δικαίωμα της ελευθερίας, της ένομης τάξης, του δικαίου αν δεν καλύπτονται αυτά υπό την έννοια της σταθερότητας, τότε η σταθερότητα είναι μία έκφραση απλώς, ε, μιας, είναι μία νεκρή έννοια που δεν έχει νόημα. Ο κύριος Μπέλτερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους καλεσμένους, τα μέλη του πάνελ. Εδώ κάθομαι, εκεί πίσω. Σας ευχαριστώ, ε, ε, αξιότιμοι για αυτό που μας είπατε. Με σε αυτό που άκουσα, ότι επέστρεψε η πολιτική ψυχιατρία. Ψυχιατρική. Τα πολιτικά ψυχιατρία. Σε άλλες χώρες έχουμε φρικτές εμπειρίε από αυτά. Θυμάμαι τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι γίνεται με την ανεξιθρησκεία στη χώρα μου στη Γκούντα υπάρχει ένα ίδρυμα που εδώ και χρόνια συνεργάζεται με διάφορες κοινότητες και από χτες άκουσα ότι οι βαπτιστές που δεν είναι εγγεγραμμένοι ε, στην ε, χώρα ε, διώκονται. Θα πρέπει να τρέχουν νυχτιάτικα για να κάνουν κρυφά λειτουργίες και μυστήρια, βαπτίσεις ε, να ε, μεταλαμβάνει ο κόσμος. Είναι πραγματικά τεράστια ε, η καταπίεση αυτή. Υποτίθεται ότι θα χτίζανε ένα ορθόδοξο καθεδρικό ναό στην πρωτεύουσα. Μετά από 30 χρόνια διαπραγματεύσεων επέτρεψαν και στην Καθολική Εκκλησία. Αλλά υπάρχουν και χριστιανικές ομολογίες ε, που δεν επιτρέπεται να έχουν το δικαίωμα ε, να συνέρχονται δημοσίως και ε, επικαλούνται και τα άρθρα του συντάγματος 145 μέχρι 154 που τους δίνει αυτή την ελευθερία. Τι γίνεται λοιπόν, ποια είναι τα πιο πρόσφατα γεγονότα και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις. Στις 20 Ιανουαρίου άκουσα ότι στο Μπαντ σε ένα διαμέρισμα έγινε έφοδος ε, συνέλαβαν πάνω από 20 πρόσωπα, τους επέβαλαν αυστηρότατα πρόστιμα ε, για να τους αφήσουν ελεύθερους. Είναι πραγματικά εξωφρενικά αυτά τα πράγματα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα των Τουρκμένων πολιτών και την ανεξιδρυσία και την ελευθερία της λατρείας στη χώρα. Ευχαριστώ. Αλέτσκης, ο κύριος Αλέτσκης, ε, για δύο λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολύ σημαντικά γεγονότα. Πρόκειται για μία χώρα με ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για μία χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και το Τουρκμενιστάν γνώρισε μία ιδιάζουσα κατάσταση μετά από την αλλαγή Προέδρου είχαμε την εντύπωση ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί, κάτι το οποίο όμως δεν συνέβη. Τώρα θα πρέπει να επιλέξουμε είτε να υπογράψουμε τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ή να το σκεφτούμε. Συμφωνώ. Θα πρέπει μεταξύ των δύο κακών να διαλέξουμε το πιο ευμενές, ας το θέσω έτσι. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη ε, Ρωσία, Κίνα, Ιράν. Όλες αυτές οι χώρες είναι βασικοί εταίροι. Δεν πρόκειται για δημοκρατικές ε, χώρες. με εξαίρεση βεβαίως στην Τουρκία. Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια χώρα επαφίεστε περισσότερο, χώρα που βρίσκεται σε υποδημοκρατικές, υποδημοκρατική εξέλιξη. Κέλαμ για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι η κυρία Χάουτολα έκανε μια πολύ καλή εισαγωγή και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους του Τουρκμενιστάν για τις πάρα πολύ πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσαν. Τι μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσο περισσότερο συμμετέχουμε εκεί, τόσο περισσότερο μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Αυτό πεδείχθη ευσεβής πόθος και είναι εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κρατούμενοι δεν μπορούν να περιμένουν χρόνια όταν ενδεχομένως αλλάξει το καθεστώς, ας πούμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον κύριο Μαχμέντοφ ότι ποτέ δεν μπορεί να αλλάξει ένα κατασταλτικό καθεστώς μέσω εμπορικών σχέσεων και μόνο. Και αυτό που μας είπε η κυρία Γκόλτστον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πιέσει αυτή τη στιγμή σε περίπτωση που βάλουμε όρους στη συμφωνία. Είμαστε υπέρ των εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μας πείσει το καθεστώς ότι ε, γίνουν πραγματικές αλλαγές στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Νικολάη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να την ακούσεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την πρωτοβουλία. Βλέπουμε και πάλι πόσο ε, σημαντικά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζω ότι οι δύο αυτοί ακτιβιστές ήταν πάντα παρόντες στις μεγάλες μάχες στο Τουρκμενιστάν. Δυστυχώς αναγκαστήκατε να εγκαταλείψετε τη χώρα σας, αλλά θεωρώ ε, ότι εμείς θα σας υποστηρίξουμε για να προωθήσετε τη δραστηριότητά σας. Ο κύριος Μαμεντόφ συμμετέχει και είναι επικεφαλής της Δημοκρατικής Τουρκμενικής Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα πρέπει και στην εξορία σας να σας υποστηρίξουμε και πιστεύω ότι αυτή η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να υποστηριχθεί. Επειδή εγώ προέρχομαι από μια πρώην κομμουνιστική χώρα, γνωρίζω πολύ καλά τις, τις πρακτικές σοβιετικού τύπου. Πρόκειται για μια πρακτική που εμείς γνωρίσαμε μέχρι το 1989 και πιστεύω, συνάδελφοι, ότι εμείς την επόμενη εβδομάδα όταν θα βρεθούμε στο Αξαμπάτ θα πρέπει να θίξουμε όλα τα ζητήματα που μας έθιξαν οι προσκεκλημένοι μας. Θα τα θέσουμε στις τουρκμενικές αρχές έτσι ώστε να μας δώσουν ορισμένες εξηγήσεις για να ανοίξει ένας επικοδομητικός διάλογος υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έλεγε ένας προσκεκλημένος και εδώ θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση ότι τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν ένα μεγάλο λάθος όταν προσπάθησαν στο Τουρκμενιστάν να ορίσουν πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το πρόθυσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Πιστεύετε ότι αν υπάρξει ένας διεθνής αποκλισμός της ε, διεθνούς κοινότητας και από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα οθήσει στη, τις τουρκμενικές αρχές να τηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι όπως μας είπατε εγκρίθηκαν νόμοι οι οποίοι όμως δεν χρησιμοποιούνται. Θεωρείτε ότι αυτός ο αποκλεισμός θα ήταν χρήσιμος. Τέλος. Ωραία. Η κυρία Γκόμες για δύο λεπτά. Έχω... Είμαι στην αντιπροσωπεία που θα πάει στο Τουρκμενιστάν την ερχόμενη εβδομάδα και σημείωσα το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ε, της κατάστασης που περιέγραψαν οι καλεσμένοι μας, απέσια, τρομακτική, φρικτή και την ε, κατάσταση που ανέφερε ο πρόσωπος της Επιτροπής, ότι είναι μια ανησυχητική κατάσταση. Αναφέρθηκε επίσης εκπρόσωπος της Επιτροπής της Κομισιόν στο διάλογο, στη σημασία του διαλόγου. Μήπως θα μπορούσε να μας αναφέρει συγκεκριμένα ένα μικρό παράδειγμα, κάτι το απειροελάχιστο έστω, στο οποίο έχει επιτευχθεί πρόοδος κάτι τέλος πάντων χειροπιαστό συγκεκριμένο για να μας εξηγήσει αυτή την ε, προσέγγιση ε, της ε, ωφελημότητας του διαλόγου και της αποτελεσματικότητας της εταιρική συμφωνίας. Και του PCA. They can in touch with Αν μπορούμε να είμαστε σε επαφή Ρωτώ λοιπόν τους καλεσμένους μας εδώ πώς μπορούν να είναι σε επαφή με τους εκπροσώπους των οργανώσεων του στο Τουρκμενιστάν και ε, σύμφωνα με αυτά που είπε η κυρία Νίκολα πιστεύουν ότι ένα μποϊκοτάζ θα είναι αποτελεσματικό και επίσης ρωτώ πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς που έχει, τους μοχλούς που έχει στα χέρια της. Θα ήθελα για πέντε λεπτά να δώσω το λόγο σε κάθε προσκεκλημένο του πάνελ μας για να μας απαντήσετε σε θέματα που, στα θέματα που εθίγησαν ανάλογα με τις ε, γνώσεις σας και τις αρμοδιότητές σας. Ο κύριος Τουκμπατούλιν. Και μετά θα δώσω το λόγο στους υπολείπους. Началось с того, что считать Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω για τη σταθερότητα, αν μπορεί να θεωρείτε σταθερό το καθεστώς. Γνωρίζετε όλοι ότι πριν από δύο-τρεις μήνες οι βόρειο-αφρικανικές χώρες θεωρούνται σταθερές. Λειτουργούσαν καλά οι νόμοι και τίποτα δεν προμείνει τα όσα συνέβησαν. Τώρα φαινομενικά είναι σταθερή η χώρα, έχει νομοθεσία το Τουρκμενιστάν. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται οι νόμοι. Ο συνάδελφός μου είπε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά και την ανεργία. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που δεν μπορεί να βρει δουλειά. Εμείς έχουμε επαφές βεβαίως με το Τουρκμενιστάν, παρακολουθούμε την κατάσταση και δημοσιεύουμε στατιστικές από τη χώρα στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε δεσμούς, έχουμε επαφές με φίλους στη χώρα. Δεχόμαστε, παίρνουμε πολλές επιστολές από αγανακτισμένους πολίτες που έχουν απευδίσει και μας ρωτάνε πότε θα κάνουμε επανάσταση επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Σας παρακαλώ, όταν θα μεταβείτε στο Τουρκμενιστάν, προτείνετε το εξής σενάριο εξελίξεων. Αν ελπίζουν στην κυβέρνηση ότι θα διατηρήσουν το status quo, θα το βρουν μπροστά τους, θα ξεχυλήσει η αγανάκτηση και ο αποτροπεσμός του κόσμου και θα εκραγεί, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες. δεν χρειάζεται να τους ζητήσετε τίποτα πιο σοβαρό. Να εφαρμόσουν τους ώμους. Του νόμου, οι οποίοι ισχύουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Σε ό,τι αφορά τη ελευθερία των θρησκειών και της λατρείας είναι τεράστιο πρόβλημα για τις ομολογίε εκείνε και τις μειονότητε που προσπαθούν να φέρουν θρησκευτική ε, πολυφωνία στη χώρα. Αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύονται οι θρησκευτικές οργανώσεις εκτός αν είναι καταχωρισμένες, επίσημες αναγνωρισμένες θρησκείες. Ακόμα και αυτές οι επίσημες και αναγνωρισμένε πατάσσονται και καταστέλλονται συστηματικά. Και μουσουλμάνοι ακτιβιστές, το γνωρίζω. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, δεν σας έδωσα παραδείγματα μουσουλμάνων ακτιβιστών που έχουν φυλακιστεί. Πεθαίνουν στι φυλακές, ε, συλλαμβάνονται οι οικογένειές τους. Πάρα πολλά παραδείγματα έχουμε και εκεί. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψει συμφωνία ε, με το Τουρκμενιστάν. Είναι μέλος του ΑΣΕ το Τουρκμενιστάν και έχει δεσμεύσει αναλάβει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα εφαρμόζουν αυτά που έχουν συμφωνήσει και ο ρυθμός και ο βαθμός είναι μηδενικός. Ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο. Ουδέποτε εφήρμοσαν τα όσα δεσμεύτηκαν θα εφαρμόσουν και σε ό,τι αφορά τι επαφέ και την επικοινωνία με του πολίτε είναι κρυπτογραφημένη. Αλλά όταν μιλώ ε, στο τηλέφωνο με τη μητέρα μου δεν μπορώ να της πω αυτά που θα ήθελα να της πω. Το ίδιο και εκείνη. Ε, Νομίζω Ε, ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ε, προσέχω γιατί προσπαθούν να με δολοφονήσουν οι αρχές του Τουρκμενιστάν, έχουν στήσει συνωμοσία και πλεκτάνει εις βάρος μου. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Κάποιος είπε να κάνει τον έλεγχο και την παρακολούθηση ο ΑΣΕ. Δεν γίνεται αυτό. Έχουν να Ασκαμπάτ ε, κάνει κάποιες αποστολές με εργαστήρια, με σεμινάρια. Και οι τουρκμενικές αρχές φοβούνται τέτοιου είδους παρακολούθηση. Δεν επιτρέπουν καν την πρόσβαση στις φυλακές. Όλα κρυπτό και παραβίστο. Παρακαλώ. Ναι, το έχετε υπόψη σας ότι τα κρύβουν όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα από όλους. Ο δόκτωρ Μάμετοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους. Πολύ βασικά ερωτήματα κάνατε για τους ακτιβιστές, τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Το είπε και ο συνάδελφός μου και ίσως εκπλαγείτε, αλλά το Τουρκμενιστάν δεν είναι μια χώρα που μπορείς να πάρεις τηλέφωνο έναν υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συζητήσεις ελεύθερα. Η επικοινωνία μας με τους ακτιβιστές εκεί είναι όλοι κρυπτογραφημένοι σε κώδικες και κρυφή. Υπάρχει ολόκληρη εκπαίδευση των αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το πώς θα επικοινωνούν. Με τρόπο κρυπτογραφημένο, ακριβώς κρυφό και μυστικό. Παράδειγμα. Μπορεί να είναι παράδοξο για, αυτά, αυτό, αλλά για να μπορέσουμε εμείς να βεβαιωθούμε ότι μπορεί να φύγει κάποιος να πάει στη Ρωσία αγωνιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να πάει στη Ρωσία για να ε, έρθει σε επαφή μαζί μας, χρειάζονται δύο μήνες προετοιμασίας. Και ε, εφευρίσκουμε μια ιστορία ότι έχει συγγενεί στη Ρωσία και τον έχουν καλέσει σε ένα γάμο ή σε ε, μια βάφτιση. Τον πάμε στη Μόσχα και εκεί το συναντούμε. Έτσι έχει κατάσταση. Έτσι εργαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Γιατί εάν τον πάρουμε τηλέφωνο αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον συλλάβουν. Ε, κάποιος φυλακίστηκε για ένα χρόνο για τον εξή λόγο, για ένα απλό τηλεφώνημα όπου του ζητούσαν να δώσει κάποιες πληροφορίες. Τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν για ένα χρόνο στη φυλακή. Και μετά από ένα χρόνο βγήκε σακάτης από τη φυλακή. Έχει χάσει την υγεία του. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην επαναλάβετε τα σφάλματα των συναδέλφων σας του ΟΗΕ και των διπλωματών. Το 1995, χωρίς καμία συζήτηση, πέρασε ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη δεχόμενη την ουδετερότητα του Τουρκμενιστάν. Δηλαδή, έτεινε χείρα βοηθεία στη χώρα η διεθνής κοινότητα χωρίς να ψάξει εάν ε, ανταποκρίνονται στις ε, υποχρεώσεις τους. Είναι αδιέξοδη αυτή η συνεργασία τα τελευταία 15 χρόνια με το Τουρκμενιστάν. Ε, ελπίσανε κάποιοι ότι ε, αυτό θα φέρει τη δημοκρατία στη χώρα. Το αντίθετο έγινε. Έχουμε ένα από τα πιο καταπιεστικά καθεστώτα, τα πιο κατασταλτικά του κόσμου. Όταν μιλάτε λοιπόν για συνεργασία με το Τουρκμενιστάν, να βασίζεται αυτή σε κάποιες προϋποθέσεις και κάποιους όρους και αυτή τη στιγμή ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις της η χώρα να αποφασίσετε αν και κατά πόσο είναι έτοιμη να ακολουθεί στο δημοκρατικό δρόμο. Εάν δεν ακολουθηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, εάν δεν γίνουν σεβαστοί οι όροι, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε συνεργασία δεν πρόκειται ποτέ η χώρα να βελτιώσει τις επιδόσεις της για το καθεστώς. Πρόκειται για ένα καθεστώς πάρα πολύ σκληρό, κοινικό, που μπορεί να σας εξαπατά και να ψεύδεται εις το διηνεκές. Και απλώς κάνετε συναντήσεις, συζητάτε και σε τελική ανάλυση δεν αλλάζει τίποτα. Και ποιος υποφελείται το καθεστώς έχουν μαζί σας επαφές. Αυτό είναι αδυναμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αποδοχή του καθεστώτος. Και παίζει το ρόλο που του επιφυλάσσει ένα τέτοιο καθεστώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ, ακούστε τις μητέρες των οποίων ε, φυλακίστηκαν σε αυτή τη χώρα. Ακούστε τις μητέρες εκείνων που, εκείνων που πέθαναν από ναρκωτικά ή τους έχουν βάλει στα μαύρα κατάστοιχα. Είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική να προσπαθείτε να φέρετε τη δημοκρατία σε μια χώρα μέσω της οικονομικής συνεργασίας και του εμπορίου. Η Βερμανία, το ίδιο παράδειγμα. Ή η Ζιμπάμπουε. Μπορεί να συζητάτε με τον Ρόμπερτ Μουγκάμπε όσο θέλετε. Αυτός δεν πρόκειται να αλλάξει. Και το ίδιο ισχύει για τον Μπέρντι Μουχαμέντοφ, τον πρόεδρο της χώρας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόλστον έχει το λόγο για πέντε λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους έθεσαν ερωτήσεις. Καταρχάς το Human Rights Watch δεν είναι εναντίον των επαφών, ούτε υποστηρίζουμε την απομόνωση της χώρας ή του καθεστώτος. Αυτό που υποστηρίζουμε είναι μία δέσμευση η οποία θα προωθήσει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί έχουμε μία ριζικά διαφορετική θέση από την Κομισιόν. Η Κομισιόν πιστεύει ότι ο διάλογος είναι καλός ε, ως αυτοσκοπός ε, εμείς έχουμε μια αντίθετη άποψη. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Είμαστε υπέρ των επαφών του διαλόγου, αλλά ο διάλογος πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και να όχι να είναι αυτός σκοπός. Έτσι έρχομαι στο, στη δεύτερη μου παρατήρηση που αναφέρεται στη δήλωση που έγινε ότι η σχέση αυτή, ο διάλογος αυτός ε, είναι μακροπρόθεσμος, έχει μια μακροπρόθεσμη εξέλιξη και δεν μπορούμε να αναμένουμε μεταρρυθμίσεις μέσα σε μια νύχτα. Βέβαια, η υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων, εξωτερικής πολιτικής, ε, ε, πρέπει να ερωτηθεί και να μας απαντήσει τι εννοείται μακροπρόθεσμα, πόσο πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αποτελέσματα διότι η εμπειρία μας για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες της Κεντρικής Ασίας και στο Τουρκμενιστάν βέβαια δείχνει ότι δεν επιτυγχάνονται αποτελέσματα εάν δεν υπάρχει έντονη εξωτερική πίεση. Οι κυβερνήσεις αυτές δεν έχουν την πολιτική βούληση για αλλαγές, οπότε ο μόνος τρόπος να σημειωθεί πρόοδος είναι εξωτερική πίεση και αναφέρομαι τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Παλέσκης ότι είναι μια δύσκολη επιλογή το να προχωρήσουμε μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας είναι βεβαίως μια επιλογή αλλά είναι δύσκολο εμείς πιστεύουμε ότι η προοπτική των αναβαθμισμένων σχέσεων μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο πρόοδου. Δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτό μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χρησιμοποιήσει το μοχλό του ενδεχόμενου αναβάθμισης των σχέσεων για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ασκηθεί, να ασκηθεί περισσότερη πίεση, να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο αυτό ε, για ορισμένες παραχωρήσεις και βελτιώσεις. Δυστυχώς έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο μοχλός πίεσης. Δεν είναι όμως ε, χαμένη η υπόθεση έχετε να αποφασίσετε αυτή τη στιγμή. Θα υπογράψετε, ή θα δεχθείτε την συμφωνία εταιρική σχέσης χωρίς ανταλλάγματα ή θα τη χρησιμοποιήσετε ως κίνητρο, ως δόλωμα αν θέλετε, για την παροχή παραχωρήσεων και για την επίτευξη κάποιας πρόοδου πριν τέλος πάντων προχωρήσει η συμφωνία αυτή. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας χρησιμοποιείται πολλές φορές για να θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε καλύτερη θέση, σε πιο δυνατή, να της δώσει ισχύ δηλαδή και δύναμη εμείς δεν βρίσκουμε αποδεικτικά στοιχεία να υποστηρίξουν αυτή τη θεωρία. Δηλαδή ότι το PCA, αυτή η εταιρική συμφωνία, ε, ενδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν. Όμως, αυτό που βλέπω εγώ να γίνεται είναι να εκδίδονται ανακοινοθέντα τύπου, να διοργανώνονται διμερείς συζητήσεις, συναντήσεις. Ε, η επίσκεψη που θα γίνει την άλλη εβδομάδα είναι μία ε, ανακοίνωση τύπου μισής σελίδας με δύο γραμμούλες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που λένε ότι η Κομισιόν τονίζει τη σημασία της πρόθεσης ε, του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εταιρικής συμφωνίας. Μα δεν είναι αρκετό αυτό. Αυτό είναι εντελώς ανεπαρκές για να προχωρήσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Αυτό, αυτή η φρασούλα, αυτές οι δύο-τρεις γραμμές δεν είναι ένα επαρκές εργαλείο για να προωθηθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σίγουρα μπορεί και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Και εδώ με το πλαίσιο της ε, ενδεχόμενης αυτής συμφωνίας παρουσιάζεται μια ιστορική ευκαιρία επιτέλους να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν. Ευχαριστώ την ε, δόκτωρα Γκόλστον. Νομίζω ότι προβλέπετε μια ε, μία απάντηση από τον κύριο Φισέρα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μέσα σε δύο λεπτά την ερώτηση της κυρίας Γκόμες, η οποία δεν έχει απαντηθεί. Ευχαριστώ. Καταγράψαμε τα διάφορα σχόλια και τις απαντήσεις σε σχέση με την ανεξιθρησκεία. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και ένα από τα ζητήματα που ε, θίξαμε στο Διάλογο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, η επόμενη σύνοδος θα γίνει τον Ιούνιο και εάν θέλει η Ευρωβουλευτής να θίξει αυτό το ζήτημα, πολύ ευχαρίστως. Μας ενδιαφέρουν οι όροι κράτησης των φυλακισμένων ιδιαίτερα. Ως προς το ερώτημα της κυρίας Γκόμες, ως ε, μέλος της ΕΙΕΔ δεν είναι να ε, παρακολουθήσω το κατά πόσο το Τουρκμενιστάν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τη δική μας πολιτική δεσμεύση ανοχαίνομαι, διότι η οργάνωση Human Rights Watch είναι υπέρ της δέσμευσης και όχι υπέρ του αποκλεισμού ή της απομόνωσης. Πιστεύουμε ότι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα και ως προς την ε, Διεθνή Εμπορική Συμφωνία δεν ε, είχαμε καιρό να την εξετάσουμε, αλλά η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα καλύτερο μέσο στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ. Bene, Ωραία. Σας ευχαριστούμε κύριε Φίσερ. Η πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κάτι να προσθέσει, η κυρία Χάουταλα. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη. Θα ήθελα να είμαι ιδιαίτερα ευγενής, αλλά με εκπλήσει η η προσέγγιση και η υπερφύαλη στάση της ΕΙΕΔ σε σχέση με το τι βλέπουμε στην χώρα. Κανένας δεν είπε ότι θέλουμε να απομονώσουμε το Τουρκμενιστάν. Όμως θέλουμε μια πολιτική δέσμευση η οποία πραγματικά να δείξει ότι υπάρχει διαφορά, ειδοποιώ διαφορά. Δεν είμαι πεπισμένη. Αντίθετα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική πολιτική θέληση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. γιατί αυτό σημαίνει ότι θα θυσιάσετε ε, ορισμένα στοιχεία τα οποία σα βρίσκουν πολύ σύμφωνους όταν προβαίνετε προς δηλώσεις, σε Νομίζω ότι αυτό το θεσμικό θέμα μεταξύ ΕΙΕΔ και Κοινοβουλίου είναι πολύ σοβαρό, διότι όταν υπάρχει νομική πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με τον μηχανισμό εποπτείας του Κοινοβουλίου που δείχνει ότι υπάρχει στρέβλωση ε, ισορροπημένης προσέγγισης, αυτό θα πρέπει να το υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο έγκαιρα. Ευχαριστούμε κυρία Χάουταλα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους εκεί ήρθαν από πολύ μακριά η κυρία Γκόλστον από τη Νέα Υόρκη και εσείς αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που φανταζόμαστε για να είσαστε εδώ μαζί μας. Η κυρία Νικολάη, η οποία τώρα δεν είναι παρούσα, η οποία συλλέγει στοιχεία πριν από την έγκριση στην Ολομέλεια της έκθεσής της και η κυρία Γκόμες που στις 26 του μηνός, στις 26 Απριλίου θα μεταβεί στο Τουρκμενιστάν, θα έχει συλλέξει διάφορα στοιχεία αξιολόγησης και αποτίμησης. Ε, εμείς ε, πλουτίσαμε από αυτή τη συνάντηση, εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας, από τις εμπειρίες σας που δεν ήταν καθόλου ευχάριστες. Ο δόκτωρ Τουμπατολίν μας είπε και μας έδωσε πολλά στοιχεία να ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κοντά σας και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας. Το επόμενο θέμα μας, μα, το επόμενο θέμα θα διεξαχθεί, θα συζητηθεί και κλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό θα ήθελα τα μέλη που έχουν άδεια να παραμείνουν, να παραμείνουν και οι άλλοι να αποχωρήσουν αμέσως. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά. Ε, Στο μεταξύ, και ενώ θα οργανώσω